8 Ιανουαρίου 2009 και σύμφωνα με το άρθρο 42 του κανονισμού 45-2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και μετά από τις διαβουλεύσεις της Επιτροπής Θεμελιωδών Ελευθεριών δέχθηκε τον διορισμό του κ. Πίτερ Χάστινγκς ως εντεταλμένου την προστασία των προσωπικών δεδομένων και του κ. Τζοβάνι Μπουταρέλη ως αναπληρωτού του. Πρόκειται για κοινό διορισμό που γίνεται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από το Συμβούλιο Υπουργών και θα υπογράψω προσωπικά την Τετάρτη μαζί με τον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου της, ε, τη σχετική απόφαση. Σας ανακοινώνω επίσης ότι στις 14 Ιανουαρίου, Τετάρτη, σύμφωνα με το άρθρο 68 του κανονισμού, θα υπογράψω έξι ε, νομοθετήματα τα οποία έχουν εγκριθεί στα πλαίσια της διαδικασίας συναποφάσεως και θα τα βρείτε στα σημερινά πρακτικά.